We will continue our meeting with... Θα περάσουμε στο σημείο 21. Σχέδιο σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σε ό,τι αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί το καθεστώ του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνοντας τον αριθμό των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου. Δεν είναι εδώ ο εισηγητής. Το ρόλο του θα αναλάβει η κυρία Ντελβό, που είναι η αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας. Έχει το λόγο, η κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είμαι εισηγητή. το πλέον το ξεκαθαρίσουμε αυτό και δεν, έχω σκοπό να γίνω εισηγήτρια. Αντικαθιστώ τον κύριο Μαρίνιο Επίντο στο μεταξύ απλώς. Καλό είναι να υπενθυμίσω ότι είμαστε σε μια διαδικασία δεύτερης ανάγνωσης και το χρονοδιάγραμμα μας πιέζει πολύ. Εάν θέλουμε να πούμε οτιδήποτε επί του θέματος, θα πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετήσουμε μια έκθεση ή κάποιες τροπολογίες, μια θέση τέλος πάντων, το αργότερο, στη δεύτερη σύνοδο του Οκτωβρίου. Αλλιώς περνάει η προθεσμία και θα περάσει η θέση του Συμβουλίου χωρίς εμείς να πούμε τίποτα. Δεν ξέρω πορτογαλικά. Δεν μπορώ να σας συνεψίσω λοιπόν την έκθεση αλλά οι τροπολογίες που παρουσίασε ο κύριος Μαρίνιο Πίντο στην έκθεσή του ε, μεταφράστηκαν σήμερα το πρωί και σήμερα τις λάβαμε στα αγγλικά. Και μπορώ λοιπόν εν συντομία να σας εξηγήσω το περιεχόμενο αυτών των ε, τροπολογιών. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες, αλλά χοντρικά ομαδοποιούνται σε έξι σημεία. Πρώτον, ο κύριος Μαρίνιο Πίντο προτείνει να διαγράψουμε στην αιτιολογική σκέψη όλες τις αναφορές στην αύξηση του όγκου εργασίας του δικαστηρίου, στι απαράδεκτες προθεσμίες, στην περιπλοκότητα των υποθέσεων, όλα αυτά που μιλούν για αύξηση της εργασίας του δικαστηρίου, θέλει να τα διαγράψουμε. Καθώς και την αιτιολογική σκέψη που λέει ότι ότι υπάρχει ανάγκη αύξησης του αριθμού των δικαστών. Αυτά για, την αιτιολογική σκέψη. Εν συνεχεία, για τα άρθρα. Προτείνει μια τροπολογία. Λέγοντας ότι το δικαστηρίο θα έχει το πολύ 40 δικαστές, αλλά όχι εν μία σε μια φορά, κάθε φορά, κάθε φορά που θα χρειάζεται επιπλέον δικαστή, το δικαστήριο θα πρέπει να δικαιολογήσει το αίτημα. Να δικαιολογήσει καλύτερα το αίτημα. Εν συνεχεία, προτείνει να έχουμε 19 επιπλέον άτομα και στη γραμματεία και στις... Ε, και προτείνει επίσης να αυξήσουμε τους μεταφραστές και αντί να έχει κάθε δικαστής τρεις βοηθούς, να έχει τέσσερις. Επίσης προτείνει τη δημιουργία μιας ειδικής επιτροπής που θα συνετέχει το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή για να εξετάζει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης. Μια άλλη τροπολογία προτείνει η Κομισιόν να τηρεί μια στάση επιτήρησης. Απέναντι σε όλα τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, όπως γίνεται από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επίσης, οι διαδικασίες διορισμού. Ο εισηγητής θα ήθελε να εμπλέξει το Κοινοβούλιο σε αυτές και προτείνει ότι το δικαίωμα διορισμού παραμένει στα κράτη-μέλη, αλλά μετά από διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν το κράτος μέλος έχει ήδη ένα άντρα δικαστή, θα πρέπει να έχει υποψήφια γυναίκα. Και αντίστροφα, εάν έχει δικαστή ήδη γυναίκα, θα πρέπει ο υποψήφιος να είναι άντρας. Για την επόμενη φορά προφανώς. Αυτές είναι οι τροπολογίες, έτσι τις κατάλαβα. Όλες οι πολιτικές ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν πιο προσεκτικά με την πρόταση. Αυτά σας τα λέω εν είδη αναπληρώτριας και αντικαστώ βέβαια τον κύριο Μαρίνιο Επίντου. Ευχαριστώ κύριε Ρέγνερ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για την παρουσίαση για το, τις τροπολογίες. Οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες θεωρώ. Ωστόσο, να σας υπενθυμίσω και το παρακάτω. Ο φάκελος αυτός είναι ένας φάκελος ο οποίος μας απασχολεί επί πολύ καιρό και έχουμε και χρονική πίεση πλέον. Για όσους ε, δεν ήταν στην τελευταία θητεία, να σας πω ότι είχαμε ψηφίσει και την ε, προηγούμενη θητεία και μετά ε, πέρασε το μπαλάκι στο Συμβούλιο. Τώρα ψήφισε λοιπόν και το Συμβούλιο και τώρα ε, το Συμβούλιο θέλει να αναφερθεί στους, στον των δικαστών στο δικαστήριο. Και στη φάση αυτή λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε και τον χρονικό παράγοντα. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα προτείνουμε από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ και άλλοι φαντάζομαι τον τελευταίο καιρό μιλήσαμε με την Λουξεμβουργενή Προεδρία και εδώ πρέπει να πούμε ότι ασχολείται εδώ και πάρα πολύ καιρό το θέμα αυτό. Και να σας πω ότι υπάρχουν ε, δεν είμαι υπέρ του να διπλασιαστούν οι δικαστές στο δικαστήριο, αλλά είμαι και ρεαλίστρια. Θέλουμε λοιπόν μια γρήγορη λύση, άμεση λύση ή θέλουμε σε κάθε περίπτωση να γίνουν μεγάλες αλλαγές σε σχέση με τις προτάσεις του Συμβουλίου. Και να καταπιαστούμε με μεγάλες διαπραγματεύσεις, μακροχρόνιες, οι οποίες έχουν τον κίνδυνο τελικά να επιβληθεί η γνώμη του Συμβουλίου. Άρα, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να η υπόψη στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για μας ως Κοινοβούλιο. Και εδώ θα συμφωνήσω με τις προτάσεις της κυρία Δελβό να υπάρχει και μια ισορροπία μεταξύ γυναικών και ανδρών δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστηρίο. Αυτό συνάδει και με τις ε, συνθήκες και πιστεύω ότι θα πρέπει να το εισαγαγεί ως στοιχείο το Κοινοβούλιο και δεν το λαμβάνει υπόψη η άποψη του Συμβουλίου. Κάτι άλλο, ότι σε κάθε περίπτωση φυσικά και είναι απαραίτητο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφαίνεται αποτελεσματικά γρήγορα προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Και φυσικά θα πρέπει να λογοδοτεί και θα πρέπει ασφαλώς να μην διαρκούν ε, πάρα πολύ οι δικαστικές αποφάσεις, οι έκδοση των αποφάσεων. Άρα, στέκει το να αυξηθεί ο ρυθμός των δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και για να ακολουθήσουμε αυτή τη ροή της σκέψης, αν όντω διπλασιάσουμε τον αριθμό των δικαστών όπως προτείνει το Συμβούλιο, θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο μια τέτοια ρύθμιση να ελεγχθεί σύντομα. Δηλαδή, να περιλαμβάνεται μια ρήτρα η οποία θα προβλέπει επακριβώς έλεγχο του κατά πόσον ο διπλασιασμός του αριθμού των δικαστών ήταν όντω εύλογος, σωστός και αποτελεσματικός. Υπό αυτούς τους όρους θεωρώ ότι θα μπορούσαμε με ρεαλιστικό τρόπο να ακολουθήσουμε την πρόταση του Συμβουλίου για να διπλασιάσουμε τον αριθμό των δικαστών, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι ενθουσιώδης η ομάδα μου για τον διπλασιασμό, αλλά πιστεύουμε ότι αποτελεί μια ρεαλιστική λύση υπό τις συνθήκες τι οποίες σα ανέφερα. Ευχαριστώ, κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι πλέον δεν βρισκόμαστε σε μια ιδανική κατάσταση, γιατί πολλοί από εμά θα θέλαμε να έχει εγκριθεί η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου, να προσθεθούν δηλαδή 12 δικαστές. Και υπάρχει και ο παράγοντας του χρόνου. Να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι θα γίνει τελικά αυτή η αλλαγή και τελικά να μην χάσουμε την δυνατότητα να δραματίσει το ρόλο του το Κοινοβούλιο όπως του αρμόζει. Πιστεύω λοιπόν ότι η γραμμή την οποία προτείνει η κυρία Ρίγνερ είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη ως πολιτικές ομάδες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία για την ανάγκη αυτής της μεταρρύθμισης. Δεν χρειάζεται να διαγράψουμε τις τροπολογίες που αφορούν την αύξηση του φόρτου του δικαστηρίου και την ανάγκη έκδοσης πιο πολλών αποφάσεων πιο γρήγορα. Άρα, υπό την έννοια αυτή δεν σύμφωνο με τον κύριο Μαρία Ντεπίντο, ο οποίο είναι ο μόνιμο εισηγητή. Νομίζω ότι είναι κατεξοχήν καθήκον μα να διασφαλίσουμε τη λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία του δικαστικού συστήματο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ αλλιώ θα πετύχουμε το κράτο δικαίου, αν δεν έχει το δικαστικό σώμα επαρκή πόρου. Είναι και θέμα χρονική συγκυρία, ξέρετε. Δύο, λοιπόν, δυνατότητες. Είτε θα ακολουθήσουμε την ε, τοποθέτηση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση και θα θέσουμε κάποιες απαιτήσει ε, για να εξολογήσουμε τις ανάγκες των δικαστών. Αλλά νομίζω ότι θα ξεκινήσει μια πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση με το Συμβούλιο για την ανάβρη... Ε, εξέβρεση και δεν θα καταλήξουμε σε καλύτερη λύση τελικά. Αυτό θεωρώ ότι είναι γεγονό. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και κάποιες αξιώσεις σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της εφαρμογή, της μεταρρύθμισης και τέλος. Έχει έρθει ο καιρό να φροντίσουμε στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει η ανάλογη εκπροσώπηση των δύο φύλων. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάνε τα πράγματα, αλλά τελικά το βασικό είναι να μην καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου θα και θα βγει από πάνω το Συμβούλιο και θα επιβάλλει διπλασιασμό των δικαστών και δεν θα έχει ακουστεί και το Κοινοβούλιο και δεν θα έχει περάσει και καμία α, ε, αξίωση τους σε ό,τι αφορά τα φύλλα κτλ. Mr. Ακόμα και αν ε, είναι αξιολογηθεί με διαφορετικό τρόπο ο διπλασιασμό των δικαστών, θέλω να σα ε, πω το εξή. Όλοι ξέρουμε ότι τα ευρωπαϊκά ε, όργανα γενικώ την χάνουν αμφισβητήσεων. Ξέρετε τη συζήτηση που γίνεται για την Ευρώπη και νομίζω ότι ένα σημαντικό κομμάτι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί καλύτερα. Να αρχίσει να λειτουργεί καλύτερα το κράτος δικαίου στην Ευρώπη. Και γι' αυτό εγώ προτιμώ και για λόγους σταθερότητας της Ευρώπης γρήγορα να καταλήξουμε σε μια ρεαλιστική λύση και αυτή την ε, πρόταση να την προωθήσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε. Τα θέματα που, τον, που είπε η κυρία Ρέγνερ επίση ε, θέλω να τα υπογραμμίσω και εγώ. Το θέμα κυρίω των ποσοστώσεων, τη κάλυψης, της από γυναίκε και άντρε. Εγώ θέλω να έχουμε μια σκληρή ποσόστοση. Αν δεν υπάρξει σαφής διαχωρισμός, σαφής κατανομή ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών θα πρέπει να κρατούνται η θέση άδεια, να μην καλύπτεται. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε σαφέστεροι, πιο οξείς και επίσης θα πρέπει να γίνει σωστή λεπτομερής ε, ανάλυση αυτών των αριθμών που προτείνεται τελικά για την κάλυψη των θέσεων των δικαστών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η Ευρωπαϊκή Ένωση διανύει μια ηθική κρίση που συνδέεται με διάφορους παράγοντες. Το πρόβλημα της μετανάστευσης που δημιουργεί διχόνηση μεταξύ των κρατών μελών και που δείχνει την αδυναμία της Ευρώπης και την απόλυτη αποτυχία για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, το πρόβλημα της Γεωργίας, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη Γαλλία, όπου η Γεωργία είναι έξαλλη αντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τους συναντήσω και προσωπικά για να μπορέσω να του καθησυχάσω αν γίνεται, την Πέμπτη και το πρόβλημα του δικαστηρίου. Το πρόβλημα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δείχνει την ηθική αυτή κρίση. Να σας υπενθυμίσω το πλαίσιο αυτής της ιστορίας. Ε, υπάρχει μια υπόνοια ε, που καταγγέλθηκε από το γαλλικό τύπο. Έτσι. Θέλω να δω τι συνέχεια δόθηκε σε αυτές τις υπόνοιες που υπάρχουν ε, που δεν μπορούμε να αφήσουμε έτσι και δεν μου δόθηκε καμία απάντηση. Ε, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα με αυτό το θεσμικό όργανο και δεν απαντάει όμως. Εδώ θέλουμε να αντιπλασιάσουμε τον αριθμό των δικαστών του δικαστηρίου. Δεν καταλαβαίνω ποιοι είναι οι λόγοι. Γιατί όπως ο εισηγητή ο κ. Μαρίνιε Πίντο και εγώ πιστεύω ότι το άχθος που βαραίνει το δικαστήριο, τα όγκος εργασίας δεν δικαιολογούν αυτά τα ριζικά μέτρα. Το Συμβούλιο προσπαθεί δια της βίας να το περάσει και αυτό δείχνει πού βάζει το Κοινοβούλιο. Εγώ για τη διαδικασία έχω δύο παράπονα. Πρώτον, στην πρώτη ανάγνωση υποτίθεται την κάναμε μάλλον, μάλιστα την, το 2011 στο, με το προηγούμενο κοινοβούλιο, στην προηγούμενη θητεία. Αλλά ήταν διαφορετικό αυτό το project από αυτό που μας εξ, ε, παρουσιάζουν σήμερα. Επομένω, υπάρχει μια καταφανή παραβίαση τη κοινοβουλευτική διαδικασία. Το δεύτερο πρόβλημα το ανακαλύπτουμε σήμερα. Ότι η έκθεση του εισηγητή που γράφεται στα πορτογαλικά δεν έχει μεταφραστεί. Είναι ενοχλητικό λοιπόν να πάρουμε θέση σε μια αμετάφραστη έκθεση. Ε, έχουμε βέβαια τι τροπολογίε στα αγγλικά, τέλο πάντων καλύτερα από το τίποτα, αλλά μόνο στα αγγλικά. Υπάρχει ένα σοβαρό το πρόβλημα διαδικασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία. Επαναλαμβάνω, είμαι πεπισμένος ότι ο διπλασιασμός του αριθμού των δικαστών δεν είναι απαραίτητος. Ακούσαμε όταν ε, στην Επιτροπή μας ε, είχαμε την ακρόαση των δικαστών, ε, οι δικαστές να μας λένε ότι δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, ότι δεν ήταν απαραίτητο. Και επομένω η λύση του κύριου Πίντο είναι απόλυτα λογική, συμφωνώ με διάφορα πράγματα από αυτά που προτείνει, τη διαγραφή, τη... στην αναφορά που γίνεται παντού το όγκο εργασία και την ανάγκη να αυξήσουμε τον αριθμό των δικαστών, ε, η ανάγκη να προσλάβουμε περισσότερους εισηγητές του δικαστηρίου ε, για να βοηθήσουν τους δικαστές να διεκπαιρέσουν τα καθήκοντά τους και μια, να δημιουργήσουμε μια επιτροπή που θα εξετάσει τη λειτουργία της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης, γιατί όχι, και να υπάρχει και μια ε, υποχρέωση σεβασμού της ισορροπίας ανδρών γυναικών. Κανένα πρόβλημα. Αλλά έχει μέχρι θα πρέπει να αποφανθούμε τώρα ή υπό την πίεση του Συμβουλίου υποχωρούμε και το αφήνουμε να κάνει ό,τι θέλει και επομένως δεν εξυπηρετούμε και τίποτα ή προσπαθούμε να υπερασπιστούμε μια λογική θέση κάτω την άποψή μας. Και αν θεωρούμε ότι υπερασπιζόμαστε μια τέτοια θέση, λογική δηλαδή, πρέπει να υπερασπιστούμε μέχρι σε σχάτων. Thank you very much, uh, Mrs. Ευχαριστούμε. Ένα σημαντικό σημείο που αναφέρει στις τροπολογίες του εισηγητή και ακούστηκε και από κάποιου από τους εμπειρογνώμονε που είχαμε για το θέμα αυτό, είναι ότι η αύξηση του αριθμού των δικαστών θα οδηγήσει σε αύξηση της αποτελεσματικότητας, αν αυξηθεί αναλογικά και το αριθμό του προσωπικού. Οπότε θα ήθελα να θέσω το ερώτημα. Αν αποφασίσουμε να αυξήσουμε, να διπλασιάσουμε τον αριθμό των δικαστών, θα θα ήμασταν έτοιμοι να ζητήσουμε και την ανάλογη αύξηση του αριθμού του προσωπικού. Γιατί είναι σημαντικό, ανεξάρτητα από την ε, απόφαση που θα λάβουμε για τον αριθμό των δικαστών, αυτή η μεταρρύθμιση να πληρεί τον στόχο για τον οποίο δημιουργείται. Να αυξηθεί δηλαδή η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα κατά την οποία λαμβάνονται οι ε, αποφάσεις του δικαστηρίου. Ε, Σα ευχαριστώ. Ε, κυρία Χάνιμπολ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι δύσκολο το θέμα. Το συζητάμε και εδώ και καιρό. Και επισκεφθήκαμε μερικοί εξημών το δικαστήριο και όλοι οι δικαστέ ήταν ξεκάθαροι ότι υπάρχουν καθυστερήσει, υπάρχει υπερβολικό φόρτο εργασία και οι πιο πολλοί από την Επιτροπή μα συμφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη να το αντιμετωπίσουμε το θέμα. Γιατί αυτό ασφαλώ υπονομεύει την αξιοπιστία του συστήματο, αν δεν λειτουργεί ε, αποτελεσματικά και αρκετά γρήγορα. Άρα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν πιστεύουμε όλα αυτά ότι θα πρέπει να το φτάσουμε μέχρι ότου δούμε την ίδια την έκθεση. Προφανώς, ε, λίγοι εξημών ε, διαβάζουμε στα πορτογαλικά. Τα αγγλικά ήταν λίγο περίεργο. Αλλά σύμφωνο ότι υπάρχει επίσης ανάγκη να επιταχυνθεί η διαδικασία. Αν σωστά κατάλαβα αυτά που είπε η κυρία Ντελβό, οι τροπολογίες μεταξύ άλλων προβλέπουν ότι θα πρέπει να είναι 40 στον αριθμό οι δικαστές κατά ανώτατο όριο στο δικαστήριο και 19 Εισηγητέ στο δικαστήριο. Δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό ε, θα πρέπει πραγματικά να συμβεί, αλλά να έχουμε σε κάθε περίπτωση επίγνωση του τι θα κοστίσει αυτό. Αυτό νομίζω ότι θα καθορίσει και τι προσδοκίε μα ε, για το κατά πόσο θα είναι πιο γρήγορο το δικαστήριο, πιο αποτελεσματικό και το καθεξής. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει ανάγκη λοιπόν δυνατότητα και ε, ανάγκη μεταρρύθμιση, αλλά χρειάζεται να τοποθετηθεί και το κοινοβούλιο. Χρειάζεται με ε, ταχεία αντίδραση, αλλά από την άλλη υπάρχει ανάγκη και χρόνου να διαβάσουμε την έκθεση και να αναλογιστούμε ποια θα είναι η τοποθέτησή μας ως Επιτροπή. κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που πρέπει να αποφανθούμε μόνο βάσει αυτών των τροπολογιών ε, χωρίς να μπορούμε να ακούσουμε τον εισηγητή και χωρίς να μπορούμε να διαβάσουμε και την εισήγησή του μεταφρασμένη στα αγγλικά. Διαβάζοντα τέλο πάντων τι τροπολογίε καταλαβαίνω την, το συμβιβασμό που προσπαθεί να πετύχει ο, συμβιβασ... ο Προσπαθεί και να καλύψει τις ανάγκες του δικαστηρίου για να γίνει πιο αποτελεσματικό και να μειωθεί ο χρόνος διεκπαιρέωση των υποθέσεων, ούτω ώστε όλη η διαδικασία να είναι πιο λογική και να λαμβάνεται και απόφαση σε πιο εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς να ζημιώνονται τα συμφέροντα των διαδίκων. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη από την άλλη και τις οικονομικές ανάγκες και περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συμβασμός λοιπόν ανάμεσα στα δύο αυτά. Ο διπλασιασμός του αριθμού των δικαστών όπως πρότεινε, του, όπως πρότεινε το Συμβούλιο είναι απαράδεκτο, κυρίως από οικονομική άποψη. Η πρόταση του εισηγητή να αυξηθούν το πολύ κατά 12 και κυρίως να αυξηθεί ο αριθμός των εισηγητών που ξέρετε ότι πολύ, πολύ καλά ότι κάνουν την περισσότερη δουλειά και είναι η μηχανή που κάνει το δικαστήριο να λειτουργεί. Ο, αυτός, αυτή η αύξηση του αριθμού των δικαστών και των εισηγητών μπορεί να διευκολύνει το έργο του δικαστηρίου και παράλληλα να μας εμποδίσει να κάνουμε υπερβολικά έξοδα. Στην επόμενη συζήτηση λοιπόν, ενδεχομένως, θα είναι και παρόν ο εισηγητής. Θα μπορούσαμε λοιπόν τότε να συζητήσουμε πιο ενδελεχώς την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Thank you as well. Uh, Ο κύριος Βιέφκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους για την ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική συζήτηση. Λυπάμαι που είναι απόν ο εισηγητή. Γιατί είμαστε στη δεύτερη ανάγνωση πια. Και η διαδικασία είχε καθοριστεί πριν από το, ε, το καλοκαιρινό διάλειμμα, την καλοκαιρινή διακοπή. Όλοι όσοι είχαμε ασχοληθεί με τη μεταρρύθμιση του δικαστηρίου είχαμε καθορίσει το χρονοδιάγραμμα και ο εισηγητής συμφώνησε. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τον Ιούλιο ο κύριος Μαρίνιο Επίντο δεν ήξερε το εκλογικό χρονοδιάγραμμα στην Πορτογαλία. Είναι θλιβερή η κατάσταση. Είναι θλιβερές οι εξέλιξεις αυτές με τον εισηγητή. Έχουμε αυτές τις ε, τροπολογίες στα πορτογαλικά και αγγλικά μόνο. Τελευταία στιγμή, στο πόδι. Παρότι είχαμε συμφωνήσει άλλα. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι η... το κείμενο αυτό βασίζεται, συνοψίζεται σε δύο αλλαγές, σε δύο τροπολογίες. Η θέση του Μαρίνιο Πίντο δεν έχει αλλάξει μέσα σε αυτή τη χρονιά, ούτε κατά διάνοια αρχικά ήταν αντίθετος με τη μεταρρύθμιση. Και τελικά είναι αντίθετος με τη μεταρρύθμιση. Δεν είναι πεπισμένος από τις στατιστικές, δεν είναι πεπισμένος από τα στοιχεία που του δώσαμε στις συνεδριάσεις μας. Ε, ήταν και μέλη του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Συστήματος και του δώσαν και αυτοί στοιχεία, αλλά δεν πίστηκε. Η μεταρρύθμιση γίνεται όχι γιατί θέλουμε να εφαρμόσουμε μια καινοφανή λαμπρή ιδέα. Είναι ανάγκη. Πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός. Και αν μεταρρυθμίσεις αυτή την οργάνωση, όταν τη μεταρρυθμίσεις τέλο πάντων, πρέπει να σκέφτεσαι με το βλέμμα στραμμένο μακριά στο μέλλον. Δεν πρέπει να είμαστε διστακτική και κοντόφορη. Η έκθεση του κ. Τάις χρειάστηκε δύο χρόνια για να εγκριθεί και εγκρίθηκε πέρυσι. Στο μεταξύ ε, άλλαξε η σύνθεση του Κοινοβουλίου και τώρα είμαστε ξανά, έχουμε ξανά το ίδιο θέμα. Όταν ε, ψηφίσαμε εμείς το 2014, δεν ξέραμε τη θέση του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο θεωρούσε ότι μπορεί να βρει ένα μόντους operandi ε, που δεν θα απαιτούσε τέτοια οξία αύξηση του αριθμού των δικαστών. Και εξού και η νέα πρόταση του Συμβουλίου. Τέλος πάντων, έχουμε επιτάπητος μια ριζική αναθεώρηση, μεταρρύθμιση του δικαστηρίου ή αλλιώς πετάμε στα σκουπίδια αυτό το έγγραφο. Αλλά αυτό είναι μεγάλη ευθύνη. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Αλλιώ, ποιο θα είναι ο υπεύθυνο, επιπλέον υπάρχει και κόστο. Ναι, φυσικά, αν διπλασιάσει τον αριθμό των δικαστών, θα το πληρώσει. Αλλά υπάρχουν και περισσότερε υποθέσει. Και μερικέ φορέ η εξέτασή του απαιτεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και εξάλλου μπορεί να υπάρχουν και πρόστιμα. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν μακροπρόθεσμα. Δεν είναι ότι εμείς υποχωρούμε στο Συμβούλιο, αλλά νομίζω ότι στην πρώτη ανάγνωση ήμασταν πολύ παθητικοί. Ποτέ δεν συζητήσαμε με το Συμβούλιο, γιατί ποτέ δεν το συναντήσαμε. Και γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Κυρία Ρέγνερ, κυρία Χάνιμπαλ, κυρία Χάουταλα, κυρία Ντελβό, τα είπατε αυτά, αλλά θέλω να το επαναλάβω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις απόψεις του. Και αν δεν σεβαστούμε την προθεσμία, το Κοινοβούλιο θα πει τίποτα στα πλαίσια του κειμένου. Ενώ θέλουμε να πούμε κάτι, έχουμε να πούμε κάτι. Άρα, το light motive που ήταν η ρήτρα αναθεώρησης, το, το light motive των προηγούμενων ομιλητών, η ρήτρα αναθεώρησης που θα επανεξετάσει τη μεταρρύθμιση για το αν θα πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση, καλή ιδέα να κάνουμε τη μεταρρύθμιση και μετά να δούμε αν είναι αποτελεσματική. Να το τσακάρουμε δηλαδή. Ε, επίσης η ισότητα ανδρών και γυναικών, πολύ σημαντική. Θα πρέπει να την προσπίσουμε. Υπάρχει και ένα τρίτο πράγμα, όμως εξίσου σημαντικό. Εδώ μιλάμε για μια διαδικασία σε δύο φάσεις. Εδώ μιλάμε για τον αριθμό των δικαστών, αλλά δεν είναι αυτή όλη η μεταρρύθμιση. Η μεταρρύθμιση είναι πολύ πιο περίπλοκη. Θα ήθελα εγώ να προσθέσω και ένα άλλο σημείο. Ας πούμε στο Κοινοβούλιο και στου υπόλοιπου. και στο δικαστήριο, ας πούμε, μια και θα είναι νέος, ένας νέος ε, πρόεδρος πολύ σύντομα, ότι ας δούμε τι μέτρα θα πάρει μετά τη μεταρρύθμιση το δικαστήριο, τόσο ώστε να χρησιμοποιείται πιο, πιο ορθολογικά οι δικαστές. Γιατί τώρα ε, υπάρχουν πολλές υποθέσεις ε, που πάνε συχνά στους ίδιους δικαστές, παρότι αυτοί έχουν ήδη πολλές ισορρευμένες. Και θα, ενώ θα μπορούσαν να πάνε κάπου αλλού. Το θέμα δεν είναι το νομικό προσωπικό, η βοηθή, η οι εισηγητέ, γιατί αυτοί δεν εκδίδουν αποφάσει. Οι δικαστέ εκδίδουν τι αποφάσει. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Δεν... Νομίζω ότι το δικαστήριο είναι ένας από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να έχει δύναμη. Δεν θα πρέπει να τιμωρηθεί οικονομικά, δεν θα πρέπει να το κολλήσουμε στον τοίχο, θα πρέπει να του δοθεί χώρος και χρήμα και χρόνος για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Συνοπτικά, αυτό που μας είπε η κυρία Ντελβό, που αρχικά προέρχεται από τον εισηγητή, είναι αρκετά αόριστο, δεν είναι ρεαλιστικό, δεν είναι καλές αυτές οι προτάσεις. δεν θα πρέπει ε, να συγκρίνουμε ας πούμε τελείως ανώμια πράγματα. Ε. Και νομίζω ότι αυτή την έκθεση τη χρησιμοποιεί ο εισηγητής για να κάνει κάτι το οποίο δεν αρμόζει στη δεύτερη ανάγνωση. Εδώ είναι η δεύτερη ανάγνωση, δεν είναι η πρώτη. Αυτά ταιριάζουν στην πρώτη ανάγνωση. Εγώ είμαι κατά των διαγραφών που εξηγούν γιατί είναι αναγκαία η μεταρρύθμιση. Και συμφωνώ με αυτούς που είπαν ότι είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά δεν θα υπάρξει καμία άλλη πρόταση επιτάπητος. Και ας συμφωνήσουμε με ό,τι θέλετε, αλλά Ας δεχτούμε το καθεστώς ε, ελέγχου μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης και την ισότητα των φύλων. Αυτά που τα είπατε κι εσείς δηλαδή, ας τα δεχτούμε. Thank you. Δεν ξέρω αν κάνω λάθο. Κύριε Άντερσον. I'm just wondering whether the... Αναρωτιέμαι Κατά πόσο είναι η διαδικασία για την εκλογή των ε, δικαστών ναι. που αναφέρεται στην ε, τροπολογία 15. Κατά πόσο αυτό ε, ενδεχομένως υπονομεύει την εξαρτησία του δικαστηρίου. Σε περίπτωση δηλαδή που πολιτικοποιηθεί η διαδικασία αυτή. Δεν διάβασα την έκθεση γιατί δεν μιλάω πορτογαλικά. Με μεγάλη ανυπομονησία περισμένα να τη διαβάσω. Και ελπίζω να το αναφέρει αυτό η, έκθεση. Και θα ήθελα να ακούσω και τι έχει να μας πει και ο εισηγητή σε ό,τι αφορά το σημαντικό ζήτημα τη ανεξαρτησίας του δικαστηρίου. Ευχαριστώ κύριε Δελβό. Ε, Θέλω να επανέλθω ή μάλλον να πάρω το λόγο για να πω δύο πράγματα που με ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως. Όχι ως αντικαταστάτρια του εισηγητή, αλλά ως αφύπαρκτο άτομο. Εγώ ασχολήθηκα πάρα πολύ με το θέμα αυτό, γιατί είμαι σκιώδης για τους σοσιαλιστές. Δύο πράγματα λοιπόν θέλω να πω. Πρώτον, πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των εισηγητών. Αναδικαστεί είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε σε όλες τις συζητήσεις. Και εγώ προσωπικά έφτασα στο συμπέρασμα ότι δεν είναι καλή ιδέα. Αυτή τη στιγμή ότι κάθε δικαστής έχει τρεις εισηγητές. Είναι ένας τρόπος εργασίας που προφανώς έχει λειτουργήσει. Ξεκινάω από την ιδέα ότι ένας δικαστής πρέπει παρόλα αυτά να διαβάζει τις εργασίες των εισηγητών του. Πρέπει να βρει το χρόνο. Και αν αυξήσουμε τον αριθμό των ε, εισηγητών αναδικαστή, υπάρχει ε, κίνδυνος ο δικαστής να μην μπορεί να παρακολουθήσει τον όγκο και όλων των ε, εισηγητών. Θα πρέπει να, ο δικαστής να λάβει τις ευθύνε του. Έχουμε μία διαδικασία διορισμού των δικαστών. Προτείνονται από τα κράτη-μέλη, αλλά περνάνε μπροστά από μία επιτροπή που τους εξετάζει, ας πούμε, τροποντινά πριν διοριστούν. Εάν κάνουν όμως τη δουλειά, όλη, όλη τη δουλειά οι εισηγητές, θα πρέπει αυτοί να εξετάζονται και όχι οι δικαστές. Γιατί αυτοί αποφασίζουν στην τελική. Τι νόημα έχει να εξετάζουμε λοιπόν τους δικαστές. Εγώ ποτέ δεν ήθελα την αύξηση του αριθμού των εισηγητών αναδικαστή. Δεύτερο θέμα το οποίο έθεσα είναι η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης εν γέννη. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δικαστήριο Έχουμε το, το Γενικό Δικαστήριο και έχουμε διάφορα δικαστήρια και έχουμε και ένα ειδικό δικαστήριο που είναι το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης. Στο παρελθόν είχαμε βρει αυτή τη λύση γιατί υπήρχε πολλή όγκο εργασία, πολλή φορτο εργασίας για το δικαστήριο. Γι' αυτό θέλαμε ειδικό δικαστήριο. Και τώρα αποφασίσαμε να καταργήσουμε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης. Σας λέω ότι του χρόνου, αν τόσο προχωρήσει το θέμα και ο φάκελος αυτό, αυτός θα πρέπει, ε, επειδή χρειάζεται νομοθετική πράξη για να καταργήσουμε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, θα πρέπει να φτάσει το θέμα ενώπιον του Κοινοβουλίου. Μήπως έχει νόημα, εγώ θεωρώ, να έχει ειδικά δικαστήρια παρά ε, ή ξέρω εγώ ένα πρωτοδικείο που μπορεί να οργανώνει ειδικέ ακροάσει. Θα μπορούσαμε στο εσωτερικό δικαστηρίο να έχουμε ειδικά σώματα δικαστικά. Και αυτό είναι πιθανό με αύξηση του αριθμού των δικαστών. Και όταν βλέπω τις υποθέσεις που είναι μπροστά στα δικαστηρία, διερωτώ μια και υπάρχουν πολύ περίπλοκες υποθέσεις, όσο ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, τα θέματα ανταγωνισμού, παράνομου ανταγωνισμού κτλ. Θα τα αποφασίζει ένα δικαστήριο. Θα ήμουν πολύ πιο ήσυχη εάν οι δικαστές δεν είχαν την πίεση να δώσουν το μεγαλύτερο αριθμό αποφάσεων ανά έτος, ούτως ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, καλό είναι να έχουν το χρόνο στη διάθεσή τους και να έχουμε ειδικά σώματα που θα εξετάζουν τις ειδικές υποθέσεις θα μαντέψετε από όλα αυτά ότι δεν συμφωνώ καθόλου με την γνώμη του εισηγητή. Απλώς στην πρώτη μου παρέμβαση προσπάθησα να είμαι πιστή στο πνεύμα του. Αυτά ευχαριστώ. Ο κύριος Βεύκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Να απαντήσω στον κύριο Άντερσον για την τροπολογία 15. Η τροπολογία 15 αντίκειται στη συνθήκη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι θεσμικό όργανο που διορίζει ή επιβεβαιώνει τους, ε, τον οποιονδήποτε Δικαστή αλλά θα πρέπει να γίνεται μια αναφορά στο άρθρο 255, 255. Το Κοινοβούλιο μπορεί να στείλει τον εκπρόσωπό του σε αυτή την Επιτροπή. Αυτή η τροπολογία είναι αντίθετη με τη συνδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ωραία. Η κυρία Δεν θέλω να μονοπολίσω το λόγο. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες πήραν θέση, εκτός από τους φιλελεύθερους που δεν εκπροσωπείται εδώ. Θεωρούμε λοιπόν ότι ξέρουμε τις θέσεις όλων. Και χωρίς να προδικάσουμε τις ε, τροπολογίες που θα υποβάλουν οι ομάδες, θεωρώ ότι η πλειοψηφία, εκτός από μία ψήφο, έτσι, θεωρούν ότι ο φόρτος εργασίας του δικαστηρίου αυξήθηκε πολύ και υπάρχει ανάγκη να αυξήσουμε τον αριθμό των δικαστών. Τώρα υπάρχουν και κάποιες άλλες αποχρώσεις. Ορισμένοι λένε ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουμε τυφλά το Συμβούλιο. Ας κάνουμε τροπολογίες. Τι αναμένουμε, τόσο ώστε να προτάξουμε τη θέση του Κοινοβουλίου για την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών και μία ρήτρα αναθεώρησης για να δούμε αν η λειτουργία της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης βελτιώθηκε με την αύξηση του αριθμού των δικαστών. Αυτά κράτησα τη συζήτηση. Για τις προθεσμίες. Ελπίζουμε καταρχάς ο εισηγητής να επανέλθει γρήγορα για να αναλάβει τα ενία και να υπερασπιστεί τη θέση του βέβαια. Να υπενθυμίσω όμως και τις προθεσμίες για τις τροπολογίες. Ναι, είναι σημαντικό να ξέρουμε το χρονοδιάγραμμα. για την έκθεση. Η γαλλική εκδοχή θα είναι διαθέσιμη στις 17 Σεπτεμβρίου. Η αγγλική στις 18. Οι υπόλοιπες γλώσσες στις 23 Σεπτεμβρίου. Οι υδροπολογίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. Μετά θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 13 Οκτωβρίου. Και επίσης στην Ολομέλεια. Τις 3 Οκτωβρίου θα υπάρξει μια ψηφοφορία. Ο κύριος Βεύκα θέλει το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αν ζητήσουμε μια ε, αναβολή της ε, προθεσμίας, ας πούμε 23 Σεπτεμβρίου μέχρι το μεσημέρι, είναι αρκετός χρόνος αυτός για να έχουμε μετάφραση των τροπολογιών και μετά είτε, στη, είτε την, την πρώτη σύνοδο του Οκτωβρίου είτε στις 8 να έχουμε μια συζήτηση ή πρέπει να τηρήσουμε αυστηρά αυτό το χρονοδιάγραμμα. Η γραμματεία λέει ότι είναι δυνατόν να υπάρξει αυτή η αναβολή. Ωραία. Οπότε ακολουθούμε την πρόταση του κυρίου Σβεύκα ως προς αυτό. Οπότε θεωρούμε ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 20, 23 ε, Σεπτεμβρίου συγγνώμη, μέχρι το μεσημέρι. Θα υπάρξει και έκτακτη συνεδρίαση, θα χρειαστεί έκτακτη συνεδρίαση στις 8 Οκτωβρίου το πρωί. Maybe, maybe few comments. Uh, Κάποια σχόλια για τα όσα είπατε, γιατί η κυρία Ντελβό έκλεισε τη συζήτηση πριν παρέμβω. Να πω ότι ο κύριος Βέφκα είπε ότι δεν συναντήσαμε το Συμβούλιο. Όντως, εν τω μεταξύ όμως εγώ έχω έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους της Προεδρίας και τους ζήτησα να υποβάλουν τη θέση του Συμβουλίου το συντομότερο δυνατόν. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Ένας από τους λόγους που τώρα δουλεύουμε με τόσο περιορισμένο χρόνο για τις συζητήσεις μας. Ε, καταλαβαίνω ότι η έκθεση προσπαθεί να είναι συνεκτική με αυτή της κυρία Στάιν. για την προσθήκη 12 δικαστών. As to the conditionality, uh, Για την αρισιμότητα, κυρία Ραγνέριχε ε, προτείνει να υιοθετήσουμε την θέση του Συμβουλίου και μετά να εξετάσουμε το κατά πόσο ήταν σωστή επιλογή η η πρόταση του εισηγητή λέει το αντίθετο. Ε, ας προτείνουμε λιγότερους δικαστέ, δικαστές, λιγότερο, μικρότερο αριθμό δικαστών και μετά να δούμε αν χρειάζεται μεγαλύτερος αριθμό δικαστών. Διαφωνώ με την κυρία Ντελβό ελαφρώς, κυρίως για τους εισηγητές και την αύξηση του αριθμού τους γιατί είναι ιδιαίτερος ε, περίπλοκες οι υποθέσεις ας πούμε ε, ανταγωνισμού που πρέπει να διεκπαιρεώσουν οι δικαστές και εκεί νομίζω ότι έχουν ε, πολύ καλό πεδίο δράσης οι συγητές. Άλλος κανείς? Ο κύριος Κάλλοτ θέλει το λόγο. Ε, merci, merci beaucoup, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν ονόματι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ευρωβουλευτές για την υποστήριξη που έδειξαν και την ανταπόκρισή τους στο αίτημα του δικαστηρίου να τους δοθεί απαραίτητη ενίσχυση για να εξακολουθήσει να λειτουργεί κανονικά και απρόσκοπτα. Κάτι τεχνικό και σημαντικό, αν επιτρέπετε. Να σας μιλήσω για κάποιες λεπτομέρειες. Μιλάμε για τη θέση του Συμβουλίου πάντα, έτσι. Και είναι φυσικό. Αλλά μην ξεχνάτε ότι η πρόταση δεν προέρχεται από το Συμβούλιο. Ε, είναι ένα αίτημα με βάση το άρθρο 280 που παρουσιάστηκε από το Δικαστήριο στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Και είναι ένα αποτέλεσμα προβληματισμού του Δικαστηρίου, ούτω ώστε να έχει τους απαραίτητους πόρους για την καλή λειτουργία του. Εσείς αποφασίζετε σήμερα στην πραγματικότητα για το μέλλον του δικαστηρίου και όχι για το μέλλον του Συμβουλίου. Ε, κάτι άλλο θα ήθελα να τονίσω. Συνέχεια, συνέχεια μιλάτε για διπλασιασμό του αριθμού των δικαστών. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 28 δικαστές και 7 στο Γενικό Δικαστήριο και 7 δικαστές στο Δικαστήριο Δημόσιας ε, Διοίκησης. 35 όλοι όλοι από τους 35 θέλουμε να πάμε στους 56. Σε 56. Μέσα σε διάφορα χρόνια. Έτσι. 12. 7 στο, και 7 στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης και 9 στο τέλος, στην τελική φάση, μέχρι το 2019. Είναι πολύ? Όχι, δεν είναι πολύ. Δεδομένου του αριθμού των υποθέσεων και δεδομένες της ποιότητας που θέλουμε να εξασφαλίσουμε. Ε, για να έχουμε ποιοτική δικαιοσύνη πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις διαδικασίες, τον αριθμό των υποθέσεων, αλλά κυρίως την ποιότητα της δικαιοσύνης αυτής καθεαυτής. Δηλαδή, οι δικαστές να έχουν την ηρεμία πνεύματος για να ασχοληθούν με τις περίπλοκες και λεπτές και δύσκολες υποθέσεις με την απαραίτητη ηρεμία. Κάθε, κάποιες ε, σημαντικές υποθέσεις ε, θα πρέπει να εξετάζονται μέσα σε σώματα δικαστικά πέντε δικαστών, όχι τρία συστηματικά όπως κάνουμε, τριών δικαστών συστηματικά όπως κάνουμε σήμερα. Φυσικά γίνεται συνέχεια λόγος για το κόστος. Το προσέχουμε. Μιλάμε για 13,5 εκατομμύρια ευρώ το 2019. 20% παραπάνω 20% παραπάνω σε σχέση με την πρόταση που παρουσίασε το δικαστήριο το 2011. Δεν διπλασιάζουν δηλαδή το κόστος, είναι 20% παραπάνω το κόστος. Ε, για μια πρόταση που έχει και την υποστήριξη του, του, της Κομισιόν και που δέχτηκε και το Συμβούλιο. Θα θέλανε και το Κοινοβούλιο να την υποστηρίξει αυτή την πρόταση. Και το τελευταίο, φυσικά είναι δική σας η νομοθετική διαδικασία και εμείς είμαστε λίγο στο περιθώριο. Αλλά αν κατάλαβα καλά, το να επανέλθουμε στη θέση που είχε εκφραστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη στιγμή της έκθεσης Stein για 12 δικαστές, αυτό είναι το να, σαν, να λέτε όχι, νιέτ, στην πρόταση του Συμβουλίου και να ακυρώσετε τη μεταρρύθμιση. Εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη μεταρρύθμιση. Κατεπηγόντως, τώρα. Και θα πρέπει το Κοινοβούλιο να λάβει τις ευθύνες του. Αν θέλει να υποστηρίξει δηλαδή το δικαστήριο που προσπαθεί να, έχει την, να αποκτήσει την απαραίτητη δύναμη για να διεκπαιρεώσει το έργο του. Και όπως είπε ο κ. Γεύκα, φυσικά με την απαραίτητη μεταρρύθμιση των διαδικασιών, των εσωτερικών διαδικασιών. Συμφωνώ απόλυτα. Φυσικά πρέπει να έχουμε διάλογο με το Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Κομισιόν για τα θέματα που ακούστηκαν. Την εκπροσώπηση και των γυναικών στα θεσμικά όργανα και τη δυνατότητα μια ρήτρα αναθεώρηση μετά από κάποιο φωνικό διάστημα, ούτω ώστε να μπορούμε να δούμε μαζί αν αυτό που κάναμε είναι σωστό ή αν θα πρέπει να ξαναδούμε τι κάναμε ή να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα. Υποστηρίξτε σας παρακαλώ το δικαστήριο, σας κάνω έκκληση. Το αξίζει το δικαστήριο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κανείς άλλος πέτει το λόγο. Μάλιστα. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς το λόγο, άρα μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό της ημερήσιας εξέταξης. Και να πούμε ότι θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου μια έκτακτη συνεδρίαση και μετά θα έχουμε τακτική συνεδρίαση στις 12 και 13 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρευρεθήκατε στη συνάντηση αυτή και σας εύχομαι καλά απόγευμα.